Der Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Αγαπητοί συνάδελφοι, η συνεδρίασή μας. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου 2009 της 5ης. Θα ήθελα εξ αριστερών μου καταρχάς να καλωσορίσω τον Κλάου Βέρετ, νέο Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να το, ευχαριστη... να το ευχηθώ